Hello. Good afternoon, ladies. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Ας περάσουμε στο τελευταίο πάνελ για απόψε, το οποίο φέρει τον τίτλο «Μια υφόρος και βιώσιμη γαλάζια οικονομία θα μειώσει την πίεση στους ωκεανούς». Θα ήθελα καταρχάς να πω ένα ευχαριστώ στην κυρία Μάισνερ για την όλη διοργάνωση όπως είπε και ο κύριος ε, Χέρτσικ από το ε, Γκέομαρ, ε, τόσο εύγλωτα, είναι πολύ σημαντικό να διατηρήσουμε τους ωκεανούς μας σε καλή κατάσταση. Και πρώτη, ναι, αυτή τη φανταστική ιδέα να δημιουργηθεί ένας ευρωπαϊκός οργανισμός ωκεανών. Ξέρετε ότι ξέρουμε περισσότερα για την επιφάνεια της Ελληνής από ότι για το βυθό των ωκεανών και θα πρέπει αυτό να αλλάξει. Θυμίζω ότι το τελευταίο αυτό πάνελ θα εστιάσει κυρίως ε, στο δυναμικό ανάπτυξης και δημιουργίας θέσεων εργασίας στην γαλάζια οικονομία, μειώνοντας ταυτόχρονα την πίεση που υφίστανται οι ωκεανοί. Όπως είπε ο κύριος Χέρτσικ, το 50% των τροφοίμων μας, της ενέργειας που καταλανώνουμε και ε, των φυσικών πόρων του μέλλοντος θα πρέπει να παράγονται από τους ωκεανούς. Θα ήθελα να προσθέσω όμως ότι υπάρχουν πολλές χώρες που βρέχονται από ωκεανούς που έχουν τεράστια ποσοστά ανεργίας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν για τους Ευρωπαίους και την πολιτική τους, την ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική, να εξασφαλίσουν ότι ε, θα υπάρχει μια συνοχή στην πολιτική ε, παντού, σε όλους τους κλάδους γαλάζιας οικονομίας. Τώρα βέβαια πώς θα συνδυαστούν όλα αυτά και θα ευθυγραμμιστούν με τρόπο επιτυχία. Αυτό είναι μεγάλη πρόκληση. Ε, ε, μειώνονται μεν οι ρυθμιστικοί φραγμοί και τα εμπόδια, αλλά ταυτόχρονα ε, δίνεται και μεγάλη χρηματοδότηση και είμαι σίγουρος ότι τα ανέφερε προηγουμένως αυτά ο Επίτροπος Μοέδας. Και αυτή η χρηματοδότηση κυρίως θα προέρχεται από τα ερευνητικά προγράμματα και τα διαρθωτικά ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδιαίτερα το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο για την Αλία και τη Θαλάσσια Πολιτική. Ε, ο παράκτιος, ο αλληλευτικός τουρισμός, η δατοκαλλιέργεια, η γαλάζια ενέργεια, οι θαλάσσιες βιοτεχνολογίες, ε, η εξόριξη του βυθού Όλα αυτά είναι τομείς που θίγονται από τις διάφορε πολιτικές και την νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και σε τούτο εδώ το πάνελ θα ασχοληθούμε με διάφορα από αυτά τα θέματα. Θα ήθελα επίσης να προσθέσω και μια ανησυχία που έχω. Γνωρίζετε όλοι ότι η Βρετανία επί δεκαετίες ήταν θαλασσοκράτηρα. Ε, και μάλιστα ε, πολλοί ε, θεωρούσαν ότι δάμαζαν τη θάλασσα. Και η νομοθεσία που έχουμε για την ωκεανογραφία και πολλά ε, από όσα αφορούν τα σημερινά ζητήματα έχουν έμπνευση βρετανική. Καλωσορίζω την κυρία ε, Έμα Ναβάρο, αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και της λέγω το, το λόγο για τέσσερα λεπτά. Ευχαριστώ πολύ. Είναι μεγάλη μου χαρά που βρισκόμαι εδώ με όλους σας. Να συγχαρώ καταρχάς και να ευχαριστήσω το Κοινοβούλιο και την Επιτροπή που μας δίνουν τη δυνατότητα να κάνουμε αυτή την συζήτηση για το μέλλον των ωκεανών που τόσο πολύ χρειαζόμαστε. Ένα μέλλον που όπως μας θύμισαν και οι προηγούμενοι ομιλητές αφορά τη ζωή όλων μας εδώ στον πλανήτη τους εξαρτάται. Πρέπει λοιπόν να δούμε πώς θα προστατεύσουμε και θα χρησιμοποιούμε ή θα εκμεταλλευόμαστε με τρόπο βιώσιμο του ωκεανού μας. Ακούσαμε σήμερα ότι οι ωκεανοί συμβάλλουν τα μάλα στην παγκόσμια οικονομία και είναι ε, και ε, μια δύναμη που παράγει και θέσεις εργασίας και καινοτομία και δίνουν οικονομικές ευκαιρίες για το μέλλον. Ξέρουμε ότι πέραν των οικονομικών νόμων οφελών οι ωκεανοί είναι καθοριστική σημασία για κρίσιμα θέματα του πλανήτη, από την ε, επιστηστική ασφάλεια, την ενέργεια, τους φυσικούς πόρους και την αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών. Όμως για να ε, εκμεταλλευτούμε το πλήρες δυναμικό των ωκεανών μας, θα πρέπει να εξασφαλίσουμε την προστασία τους. Πρέπει την υγεία τους να την κοιτάξουμε γιατί κινδυνεύει πολύ. Η εικόνα είναι ζωφερή και πραγματικά ε, πρέπει να κρούσουμε τον κόδωνα του κινδύνου τώρα, αμέσως. Χρειάζεται μια υπεύθυνη και βιώσιμη προσέγγιση για την οικονομική ανάπτυξη των ωκεανών, για να βεβαιωθούμε ότι ο μεγαλύτερος φυσικός πόρος του πλανήτη παραμένει ζωντανός και από αυτόν μπορούν να ωφεληθούν και να αποφεληθούν οι ερχόμενες γενιές μια βιώσιμη γαλάζια ατζέντα είναι απαραίτητη. Τα βήματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να προωθήσουν αυτή την ατζέντα είναι ευπρόσδεκτα από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, το να προωθήσουμε με τέτοια γαλάζια οικονομία που να είναι βιώσιμη, είναι προτεραιότητα. Είναι λογικό και αυτονόητο, διότι εφόσον υποστηρίξουμε την βιώσιμη ανάπτυξη και την αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών, και αυτά είναι στον πυρήνα τη δράση μα, έρχεται μαζί και η γαλάζια οικονομία. Ε, Ω μπούσουλα έχουμε ακολουθήσει φιλόδοξου κλιματικού στόχου. Ε, τουλάχιστον 25% των ε, μα, ε, τη χρηματοδότησή μα ετησίω έχει να κάνει με την κλιματική δράση. Πέρσι έφτασε τα 16 δις ευρώ. Επίσης, θέλουμε να προσφέρουμε 100 δις δολάρια για κλιματικά προγράμματα παγκοσμίω και ε, θέλουμε να έχουμε εδώ πρωταγωνιστικό ρόλο. Στη διάρκεια του χρόνου είμαστε ένα κέρια σημασία επενδυτή για την οικονομία των ωκεανών, κινητοποιώντα το κεφάλαιο του ιδιωτικού τομέα προ τους βιώσιμους στόχους και την επιδίωξή τους και στην Ευρώπη και εκτός. Ένα καλό παράδειγμα είναι το πρόγραμμά μας για την ανάπτυξη των ε, γαλάζιων ακτών στην Ευρώπη. Έχουμε αναπτύξει πολλές δυνατότητες με επενδύσεις άνω των 3,6 εκατομμυρίων ευρώ τα τελευταία πέντε χρόνια και θα συνεχίσουμε να ε, στηρίζουμε αυτόν τον τομέα σε ανάπτυξη. Επίσης η προστασία των ακτών αυτών έχει να κάνει και με το πρασίνισμα του τομέα της ναυτιλίας που είναι ένα άλλο καλό παράδειγμα. Εργαζόμαστε για την προστασία των ωκεανών από την ρήπανση από τα πλαστικά, έναν από τους μια από τις μεγαλύτερες απειλές για τα οικοσυστήματα πλέον. Γι' αυτό πέρσι μαζί με τις γαλλικές και γερμανικές τράπεζες επενδύσεων εγκαινιάσαμε την πρωτοβουλία για τους καθαρούς ωκεανούς. Τα ερχόμενα πέντε χρόνια θα προσφέρουμε δύο δις ευρώ για προγράμματα που θα αντιμετωπίσουν την αποκομιδή απορριμμάτων στους ωκεανούς, δηλαδή τα αστικά λίματα που δεν έχουν τύχει επεξεργασία και τα πλαστικά. Γι' αυτό πρέπει να ασχοληθούμε με αυτό το πρόγραμμα σοβαρά που έχει τεράστια κοινωνική εμβέλεια. Ε, όμως η ανάπτυξη της γαλάζιας οικονομίας δεν έχει να κάνει μόνο με λεφτά και χρήμα, έχει να κάνει με την ενθάρρυνση της καινοτομία και την άρση των φραγμών για νέα προγράμματα. Η γαλάζια οικονομία και τα προγράμματά της ε, μπορούν να αντιμετωπίσουν αντιμετωπίσουν δυσκολίες στην πρόσβαση στα ιδιωτικά κεφάλαια διότι πολλές φορές έχουν να κάνουν με τεχνολογικές λύσεις που είναι τελείως καινοτόμες ή με άγνωστες αγορές. Γι' αυτό με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβλέψαμε χρηματοδοτικά εργαλεία για να μειώσουμε τον κίνδυνο αυτών των προγραμμάτων και να προσελκύσουμε ιδιωτικού επενδυτέ. Αυτό είναι καθοριστική σημασία, γιατί η καινοτομία και η επιστήμη είναι κρίσιμε σημασίε για να αντιμετωπίσουμε τα θέματα της βιωσιμότητα. που ε, έχουν να κάνουν με την ε, περαιτέρω ανάπτυξη και την προστασία των ωκεανών. Όμω για να ανθίσει η γαλάζια οικονομία πρέπει να εντείνουμε την ε, χρηματοδότηση. Οι ανάγκε χρηματοδότηση είναι προφανώ πέραν των κρατικών συλλογισμών. Θα πρέπει ο ιδιωτικό τομέα να ανασκουμποθεί και να έρθει να συμμετάσχει. θα πρέπει η δική του συμβολή να ληφθούν υπόψη στις ανάλογε αποφάσει. μας. Μόνο τότε θα μπορέσουμε να κινητοποιήσουμε τι βιώσιμε επενδύσει για του ωκεανού μα για να καθοδηγήσουμε τους επενδυτές προς τη βιωσιμότητα και την βιώσιμη γαλάζια οικονομία θα πρέπει να εφαρμόσουμε τις αρχές της. Ένα παγκόσμιο πλαίσιο για την βιώσιμη χρηματοδότηση των ωκεανών που αναπτύξαμε από κοινό με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το το ΒΒΕΦ και την, το Ίδρυμα για τους βιώσιμους πόρους είναι μια αρχή. Φέτος οι αρχές αυτές θα βρεθούν στην καρδιά μιας νέας πρωτοβουλίας υπό την αιγίδα του Οργανισμού Περιβάλλοντος του ΙΕ. Αυτό ξεκίνησε ε, ως μια πρωτοβουλία 12 θεσμών και τώρα γίνεται ο κατεξοχήν κανόνας για την ε, επένδυση στους καθαρούς ωκεανούς με τρόπο βιώσιμο. Όμως ο χρόνος περνάει και έχουμε ακόμα πολλές προκλήσεις να αντιμετωπίσουμε. Προκλήσεις που θα απαιτήσουν δράση ε, συνδυασμένη και πολυμερή, αλλά και ατομικές πρωτοβουλίες όλων μας. Υπ' αυτήν την έννοια, η σημερινή εκδήλωση είναι μια μοναδική ευκαιρία για να προβάλλουμε ιδέες και να δούμε πώς μπορούμε να λάβουμε ευθύνη για την εξέβρεση λύσεων για αυτές τις προκλήσεις. Σας διαβεβαιώ ότι η ΕΤΕ παραμένει πλήρως δεσμευμένη στον αγώνα της προώθησης της γαλάζιας οικονομίας που θα κινητοποιήσει ιδιωτικά κεφάλαια και για την σύναψη εταιρικών σχέσεων με άλλου προκειμένου να υπάρξει πρόσβαση σε αυτά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ την κυρία Ναβάρο. Και τώρα θα ζητήσω από τον κύριο Πιέρ τον αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Αγοράς, Βιομηχανίας, Επιχειρηματικότητας και Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις, να πάρει το λόγο. Για τέσσερα λεπτά παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πολύ μεγάλος τίτλος για μια γενική διεύθυνση. Θα συνοψίσω με λίγα λόγια αυτά που θέλω να πω το Sky, το Copernicus, ε, ε, και η Αρκτική. Ο Ρενός είναι ένας, ένα όριο, αλλά αποτελεί ε, και ένα εργαλείο για να παρακολουθήσουμε τι συμβαίνει στη γη. Και το είπε και ο Πρόεδρος Σταγιάννη, ότι μαζί με το Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος μπορούμε να παρακολουθήσουμε μέσω του Κοπέρνικου τι συμβαίνει στη Γη. Το Κοπέρνικος είναι ένα σύστημα δορυφόρων που βασικά παρακολουθεί τον πλανήτη και παίρνει φωτογραφίες και μας δίνει φωτογραφίες για τις διάφορες καταστάσεις του πλανήτη. Στο πλαίσιο αυτό, φυσικά, οι ωκεανοί είναι πολύ σημαντικό μέρος της παρατήρησης που υλοποιούμε με το Κοπέρνικος και θα πρέπει να συνειδητοποιήσετε ότι το Κοπέρνικους ε, αξιολογείται από όλου, ακόμη και από τη ΣΥΠΑ, ως το καλύτερο σύστημα παγκοσμίω. Έτσι λοιπόν, ε, ως Ευρωπαίοι μπορέσαμε να ε, συνάψουμε ένα σύστημα, να δημιουργήσουμε ένα σύστημα που είναι το καλύτερο για την παρατήρηση της γης. Τι κάνουμε τώρα με τις εικόνες που παίρνουμε από το να αναπτύσσουμε υπηρεσίες που παρακολουθούν επίσης τι συμβαίνει στους ωκεανούς. Έτσι λοιπόν έχουμε αναπτύξει την θαλάσσια υπηρεσία που μας δίνει κάποιες προβλέψεις για τους ωκεανούς και πληροφορίες για το κλίμα στους ωκεανούς και επίσης ε, μέσω των ε, δορυφόρων μπορούμε να έχουμε μία έκθεση σε θέματα που αφορούν ε, την αύξηση του επίπεδου των υδάτων στη θάλασσα ή το λιώσιμο των πάγων. Μία άλλη πολύ σημαντική πτυχή και συνιστόσα του Κοπέρνικου είναι η παρατήρηση ε, στη θάλασσα. Χρησιμοποιείται για να παρακολουθούμε όλες τις δραστηριότητες του ωκεανού, παραδείγματος χάρη τα σκάφη στην ανοιχτή θάλασσα που βρίσκονται και τι κάνουν. Αλλά και κάτι πολύ σημαντικό να ανοιχνεύουμε τη ρήπανση και να μπορούμε να αντιδράμε γρήγορα. Μία άλλη πολύ σημαντική, σημαντική υπηρεσία είναι η υπηρεσία εκτακτής ανάγκης. Χρησιμοποιείται όταν έχουμε μία κατάσταση κρίσης, το χάρη στη Μεσανδίκη, όταν έχουμε πλημμύρες, παρακολουθεί την κατάσταση του Κοπέρνικους και μπορούμε να, μπορεί να μας βοηθήσει για να βοηθήσουμε και να σώσουμε τους ανθρώπους επί τόπου. Χρησιμοποιείται δυστυχώς σε τακτική βάση και θέλω να αναφέρω τον Δίας. Το Κοπέρνικους είναι ο μεγαλύτερος πάροχος δεδομένων στον κόσμο. Έτσι λοιπόν όλες ε, οι εικόνες, φωτογραφίες ε, που παίρνουμε μέσω του Κοπέρνικους είναι δωρεάν για όλους. Αλλά η δυσκολία είναι ότι επειδή υπάρχουν τόσα πολλά δεδομένα και ακόμη και αν είναι δωρεάν, είναι δύσκολη η επεξεργασία όλων αυτών των δεδομένων. Τι κάναμε λοιπόν ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αποφασίσαμε να πληρώσουμε ιδιωτικούς ε, παραγωγούς και να δημιουργήσουν ηλεκτρονικές πλατφόρμες με όλα αυτά τα δεδομένα. Ε, και ε, όλα τα δεδομένα διατίθεται δωρεάν σε όλους. Έτσι λοιπόν και είναι η ιδέα η ιδέα πίσω από αυτό είναι ότι όλοι θα έχουν την ευκαιρία να εξετάσουν αυτά τα δεδομένα και να αναπτύξουν υπηρεσίες και λύσεις, προϊόντα βάσει αυτών των εικόνων. Έτσι λοιπόν, αν δεν ξέρεις πια τι να κάνεις, ε, Κυριακή βράδυ βρέχει στις Βρυξέλλες, ε, πας στον Τάιας, είναι δωρεάν και δημιουργεί ε, κάτι, μπορεί να παρακολουθήσει τι συμβαίνει στον ωκεανό. Το παρουσιάζω ω αστείο, αλλά αυτό είναι ο στόχο. Ο στόχο είναι βασικά να διασφαλίσουμε ότι χρησιμοποιούνται, ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν αυτά τα δεδομένα από όλου ε, και στην Ευρώπη βέβαια και ότι αναπτύσσουμε υπηρεσίε ε, που μα βοηθούν να παρακολουθήσουμε την κατάσταση και στου ωκεανού. Και τέλο ε, Αρκτική. Γιατί αναφέρω την Αρκτική. Γιατί ακόμη ΕΝ και το Κοπέρνικους είναι ένα πολύ επιτυχές πρόγραμμα, πρέπει να το συνεχίσουμε, να το αναπτύξουμε και να το συντηρήσουμε στο μέλλον. Και τώρα, ε, στα πλαίσια τη διαπραγμάτευση του πολιτού δημοσιονομικού πλαισίου, διαπραγματευόμαστε με το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο ένα νέο διαστημικό πρόγραμμα για το μέλλον. Και ένα από τα στοιχεία που θέλουμε να αναπτύξουμε στο Κοπέρνικου, αν έχουμε υποστήριξη φυσικά από τα κράτη-μέλη και το Κοινοβούλιο, είναι η λεγόμενη Αρκτική Αποστολή. Τι θέλουμε να κάνουμε, να χρησιμοποιήσουμε το Κοπέρνικου για να παρακολουθήσουμε την κατάσταση στην Αρκτική. Γιατί ξέρουμε ότι η κατάσταση στην ε, Αρκτική επηρεάζει πάρα πολύ το κλίμα παγκοσμίω, ε, αλλά και στου ωκεανού. Και πιστεύουμε ότι θα πρέπει να έχουμε τέτοιες αποστολές, θέλουμε να τις αναπτύξουμε χρησιμοποιώντας ε, τους δορυφόρους. Και επίσης ε, θέλουμε να αναπτύξουμε μια αποστολή για την κλιματική αλλαγή. Θέλουμε να παρακολουθούμε τις εκπομπές διεξουδίου του άνθρακα. Και πάλι, αν θες να το κάνεις, το καλύτερο εργαλείο διαθέσιμο είναι το διάστημα. Έτσι λοιπόν, κάποιε φορέ παραπονιόμαστε ότι δεν είναι σχετική θέση θέση Ευρώπη σε πολλού τομεί, αλλά μπορώ να σα πω ότι με το Κοπέρνικο έχουμε ένα εργαλείο ιδιαίτερα ισχυρό. Είναι εξαιρετικό και επίσης θα είναι ένα ισχυρό μέσο για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα στους ωκεανούς. Ευχαριστώ. Uh, Ευχαριστώ πολύ, ε, κύριε Δερζού. Σε μία πρόταση, όταν μιλάτε για τον Κοπέρνικο, έχουμε την εντύπωση ότι έχει επιτευχθεί αυτό που πρότεινε ο κύριος Χέρτσικ τι λέτε για τη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Οργανισμού Θαλασσών και Ωκεανών. Μα έχουμε ε, τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος που τον ανέφερα. Γιατί να μην κάνουμε κάτι αντίστοιχο για τους ωκεανούς. Ωραία, το σημειώνουμε και μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε ότι δεσμεύεται ένας ε, υψηλός αξιωματούχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο σε κάποιους συναδέλφους μας, η κυρία Ισάσκου Πιλπάου Παραντίκα από την Άλτε, για τρία λεπτά. Η κυρία Πιλπάου Παραντίκα. Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα σας σε όλες και όλους. Καλησπέρα και ευχαριστώ ε, τους επισκέπτες, αλλά και εκείνους που διοργάνωσαν ε, αυτή την εκδήλωση όπως η Γκέινέ Μάισνερ που είναι τόσο ερωτευμένη όπως πάντα με τους ωκεανούς. Η στρατηγική αυτή η γαλάζια που αναλύουμε σήμερα είναι από τις πιο ενδιαφέρουσες χειροπιαστές δράσης του μοντέλου 2020. Από την ανακοίνωση Ευρωπαϊκής Επιτροπής το 2012 σήμανε σημαντική και οριστική αλλαγή της σχέσης μας με τη θάλασσα. Μια μετατροπή των παραδοσιακών ε, δραστηριοτήτων, διαφοροποίηση των πηγών εισοδήματο, δημιουργία νέων δραστηριοτήτων, και εκμετάλλευση της ενέργειας στη θάλασσα. Όλα αυτά βασίζονται στη βιωσιμότητα. Αναπτύσσουμε ε, την οικονομία μας μειώνοντας την πίεση στη θάλασσα. Και αυτό είναι προς όφελος των παράκτιων ε, κοινοτήτων. Για να γίνει αυτό θα πρέπει να γνωρίζουμε, ε, να παρακολουθούμε και να οργανώνουμε την προσπάθειά μας. Ε, οι παραδοσιακές δραστηριότητες τώρα βασίζονται ε, σε πολύ αυστηρές εκθέσεις ε, για τα αποθέματα. Έχουν βελτιωθεί τα αλευτικά εργαλεία και οι τεχνικές. Αναπτύσσεται η υδατοκαλλιέργεια και μετατρέπονται οι στόλοι και ο αλευτικός και ο εμπορικός. Ξεφεύγουμε από το διοξίδιο του άνθρακα. Προχωρούμε στην αυτόνομη πλοήγηση. Έχουμε ευκαιρίες για τα ναυπηγεία που είναι παραδοσιακή δραστηριότητα. Η γνώση επίση οδηγεί και σε καινοτομία και σε νέα προϊόντα και δραστηριότητε. Ε, και μπορούμε να μετατρέψουμε τις απειλέ, όπως είναι η ρήπανση από τα πλαστικά σε ευκαιρίε και στη στεριά με νέε δραστηριότητε και προϊόντα ε, για υποκατάσταση αυτών των ρηπαντών και άλλες ε, δραστηριότητες στη θάλασσα με τεχνικές καθαρισμού και συλλογής που ήδη δίνουν καρπούς. Αϊφόρος εκμετάλλευση λοιπόν ε, ενός μεγάλου θαλάσσιου πόρου που είναι η ενέργεια. Εγώ ως Βάσκα είμαι πολύ περήφανη που η μικρή μας χώρα είναι πρωτοπόρα στην έρευνα για την ενέργεια από τις παλήριες. Στο Μουτρίκου καταφέραμε να ε, παράξουμε 1,3 γιγαβάτ ε, ώρες ε, το 2016, συνδεδεμένα στο δίκτυο. Αυτό μπορεί να είναι χαμηλή παραγωγή, αλλά κανένα άλλο εργοστάσιο που χρησιμοποιεί την ενέργεια από τις παλήριες δεν το έχει καταφέρει. Χρησιμοποιεί και δοκιμάζει νέα μοντέλα μηχανών ε, έτσι ώστε ε, να ε, εκμεταλλευτεί αυτή την ενέργεια. Το ίδιο ισχύει και για τις Κανάρια, τη Κανάρια νησιά με την αιωλική ενέργεια. Άλλο κλειδί για τη στρατηγική μας είναι η οργάνωση των νέων δραστηριοτήτων. Έτσι μειώνονται συγκρούσεις και δημιουργούνται συνέργειες με την εφή εξειδίκευση ή την εγκύτητα. Και τέλος η παρακολούθηση και επιτήρηση ε, κλείνει αυτό τον κύκλο για να ε, μπορούμε να ελέγχουμε αυτές τις πρακτικές και τις αποκλίνουσες πρακτικές από αυτό το αηφόρο και βιώσιμο μοντέλο στις νέες πολιτικές μας. Γι' αυτό χαιρετίζω αυτή τη διάσκεψη υψηλού επίπεδου, έτσι ώστε να εδρεωθεί αυτή η σημαντική εξέλιξη της σχέσης μας με τη θάλασσα. Και το λέω ως Ευρωβουλευτής, αλλά και ως μέλος μιας κοινότητας, μιας κοινωνίας που έζησε, ζει και φιλοδοξεί να συνεχεί να ζει από τη γαλάζια οικονομία και που έχει ζήσει από πρώτο χέρι τι σημαίνει αηφορία και βιωσιμότητα. Γι' αυτό σας παίρνω ένα μήνυμα από την ακτή. Σε όλη αυτή την προσπάθεια μετασχηματισμού, αυτέ οι τοπικές κοινωνίες, οι παράκτιες, θα πρέπει να πρωταγωνιστήσουν. Η συμμετοχή του, είναι εκ των όνου κάνευ, έτσι ώστε αυτή η αλλαγή να προοδεύσει και να εκμεταλλευτούμε και να αξιοποιήσουμε αιώνες γνώσεων και συμβίωσης με τη θάλασσα. Και αυτές οι πολιτικές θα πρέπει να αποδίδουν στα μέλη τους ευκαιρίες, υπηρεσίες και αναγνώριση για την προσπάθεια που κάνουν έτσι ώστε να πρωταγωνιστούν σε αυτή τη βελτιωμένη σχέση με τη θάλασσα. Ε, Mar, που είναι η θάλασσα στα ισπανικά, αλλά Λαμάρ στο θηλυκό, τη λένε οι άνθρωποι της θάλασσας. Σας ευχαριστώ πολύ. Η επόμενη συνάδελφος είναι η Κλάρια Ουτζίνα Αγγιλέρα Γκαρσία από τους Σοσιαλιστές και Δημοκράτες για τρία λεπτά. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Καλησπέρα σε όλους. Έχουμε μια καλή συζήτηση, πάρα πολύ ενδιαφέρουσα σήμερα το απόγευμα. Σε αυτό το πάνελ θα ήθελα να αναφέρω κάποιες σκέψεις για να δώσω στη συζήτηση. Η γαλάζια οικονομία δεν μπορεί να αποτελέσει μόνο μια απλή έννοια ακόμη. Όταν πριν χρόνια αρχίσαμε να μιλάμε για τη βιωσιμότητα, όλα ήταν βιώσιμα. Αυτό που συνεισέφερε στη βιωσιμότητα και αυτό που δεν συνεισέφερε, αλλά όλα έφεραν την ετικέτα βιωσιμότητα. Προσοχή. Ο κίνδυνος της γαλάσιας οικονομίας είναι να γίνει μια έννοια που να καλύπτει τα πάντα. Όλα τα και, κάθε τι καινούριο. Κάθε τι καινούριο πρέπει να είναι διαφορετικό. Γι' αυτό εγώ νομίζω ότι υπάρχουν ε, κάποια στοιχεία που θα πρέπει να κάνουν τη διαφορά. Δεν μπορούμε να κάνουμε τα πράγματα όπως τα κάναμε πάντα. Θα πρέπει να δρούμε και με διαφορετικό τρόπο. Θα πρέπει να εφαρμόσουμε αυτή την οπτική για στην πράξη. Και σε σχέση και με την η κυρία Ναβάρο, θα πρέπει να αλλάξουμε και τον τρόπο με τον οποίο χειριζόμαστε τις επενδύσεις μας, ε, ιδιωτικές και δημόσιες, για να ευνοήσουμε και να προωθήσουμε αυτή τη γαλάζια οικονομία. Αυτό είναι σαφές. Μπορούμε να έχουμε τους ίδιους στόχους ή παρόμοιους στόχους, αλλά θα πρέπει να πράττουμε με διαφορετικό τρόπο και να έχουμε ξεκάθαρα πού κατευθύνουμε τις επενδύσεις μας, ιδιαίτερα τις δημόσιες αλλά και τις ιδιωτικές. Οι ωκεανοί περιλαμβάνουν τεράστιο πλούτο σε πόρους και έχουν μια τεράστια δυναμική για να προωθήσουν την οικονομική ανάπτυξη, την κοινωνία και την απασχόληση. Αν και είναι τεράστιο το δυναμικό τους, υπόκειται σε υπερβολικές πιέσεις υπερβολική εκμετάλλευση των πόρων τους, ρήπανση, αυξανόμενη βιοπικιλότητα και κλιματική αλλαγή. Όλο αυτό, όλο αυτό το μεγάλο δυναμικό μπορεί να καταλήξει διαφορετικά. Γι' αυτό πρέπει να αλλάξουμε τους τρόπους δράσης. Εγώ νομίζω ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση που θέλω να αναφερθώ, πολλοί απόψε αναφέρθηκαν και στα πλαστικά και στη ρήπανση των ωκεανών. Εγώ θέλω να μιλήσω για την ελευτική δραστηριότητα. Η τομεακή πολιτική της Ελίας, της, ε, η κοινοτική πολιτική, έφερε μεγάλες αλλαγές. Ίσως να μην ε, το αξιολογούμε επαρκώς. Γιατί μένουν πάρα πολλά πράγματα που πρέπει να γίνουν. Όμως έχουμε εγκρίνει σχέδια διαχείρισης ε, των ελευτικών πόρων ε, στα πλαίσια της κοινή ελευτικής πολιτικής και ε, για τη Δυτική Μεσόγειο αλλά και στον Ατλαντικό, στα δυτικά ύδατα όπως και στη Βαλτική ή στη Βόρεια Θάλασσα. Απομένουν πράγματα που πρέπει να γίνουν, αλλά γίνονται ήδη πράγματα για καλύτερη εκμετάλλευση και κατάργηση της υπερελίας. Και επίσης υπάρχουν μεγάλες θυσίες που γίνονται από όλους τους κλάδους. Κατά την άποψή μου, νομίζω ότι υπάρχουν κάποιες αρχές ε, που θα ήθελα να καταθέσω εδώ στη συζήτηση. Κάποιες αρχές ε, που είναι απαραίτητες ε, για αυτή την βιώσιμη γαλαζία οικονομία. Καταρχήν, για να την υλοποιήσουμε τη γαλαζική οικονομία θα πρέπει να έχουμε τη συμμετοχή και τη δέσμευση όλων των ενδιαφερομένων μερών στους ωκεανούς. Όλων. Κανένας δεν πρέπει να αποκλείεται θα πρέπει να δεσμευτούμε και να εμπλέξουμε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο για τη λήψη αποφάσεων για τη βιώσιμη γαλλική οικονομία. Δεύτερον, να έχουμε κατά νου κάτι που χρησιμοποιούμε πολύ, αλλά ενίοτε με αντιφατικό τρόπο. Την ε, υποστήριξη, τη στήριξη της καλύτερης δυνατής παροχής συμβουλών. Δηλαδή, να αξιολογούμε με τον κατάλληλο τρόπο την αξία των επιστημονικών αναλύσεων. Γιατί πολλές ε, φορές αν ε, δεν μας κάνει για την εθέτηση μιας θέσης, την απορρίπτουμε. Και το βλέπουμε εδώ και στο Κοινοβούλιο. Η επιστημονική αξία ε, των υποδοτήσεων είναι πάρα πολύ σημαντικό για την εφαρμογή της γαλάζιας οικονομίας. Και τρίτον, θα πρέπει να έχουμε κατά νου όλες τις πτυχές της βιωσιμότητας οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική πτυχή. Και τις τρεις. Αν ξεχάσουμε μία εξ αυτών, τότε δεν θα τα κάνουμε καλά τα πράγματα. Και τα τρία είναι σημαντικά για την ανάπτυξη ενός καλύτερου μέλλοντος σε ό,τι αφορά την περιβαλλοντική πτυχή, την κοινωνική και την, περιβαλλον... και την οικονομική, με συγχωρείτε. Κανένα δεν θα πρέπει να μείνει εκτός. Εγώ νομίζω λοιπόν ότι η γαλάζια οικονομία προσφέρει πολλές ευκαιρίες. Όμως θα πρέπει να ξέρουμε πού θα την κατευθύνουμε και ποιοι είναι οι στόχοι που θέλουμε να υλοποιήσουμε. Εγώ πιστεύω λοιπόν ότι θα πρέπει να συμμετέχουμε σε αυτή τη μεγάλη ευκαιρία. Όλοι θα πρέπει να συμμετέχουν. Αυτές είναι κάποιες σκέψεις που θα ήθελα να σας καταθέσω εδώ σήμερα. Βλέπουμε πολύ μεγάλες αλλαγές και δεν ε, θα ήθελα να ε, ξεχάσουμε την πρόταση να υπάρχει μια νέα υπηρεσία για τους ωκεανούς. Εμένα πολύ καλή μου φαίνεται, αλλά ξέρετε τι σκέφτεται το Συμβούλιο. Λιγότεροι πόροι για όλες τις πολιτικές για το επόμενο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Για να δούμε πώς θα κάνουμε περισσότερα, πώς θα έχουμε περισσότερα εργαλεία και μέσα με λιγότερους πόρους. Έτσι λοιπόν θα πρέπει τους πόρους που έχουμε να τους χρησιμοποιήσουμε και να τους κατευθύνουμε καλύτερα. Δεν μας διευκολύνουν βέβαια τη ζωή, αλλά νομίζω ότι είναι καλή ιδέα. Ευχαριστώ πολύ. Now I would like to... Ευχαριστώ. Και θα ζητήσω τώρα την κυρία Τομά από τους Σοσιαλιστές και Δημοκράτες να παρέμβει για τρία λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα μιλήσω γαλλικά. Θα ήθελα να πω αν ήμουν ωκεανός σήμερα το απόγευμα και έβλεπα τόσοι πολλοί να σκύβουν πάνω από το λίκνο θα ανησυχούσα. Τόσες επενδύσεις και θα έλεγα πω πω λιγάκι μαζευτείτε. Είναι σαν να παρουσιάζεται ένα νέο Ελντοράντο για πολλούς επενδυτές. Και υπάρχουν αρκετοί καλοί λόγοι. Καλοί λόγοι υπόθηκαν, δεν θα τους επαναλάβω το δυναμικό για την ανανεώσιμη ενέργεια από τη θάλασσα, το δυναμικό για τη ρομποτική που επιτρέπει να πάμε και να αντλήσουμε σε εκατοντάδες χιλιόμετρα κάτω από τη στάθμη. Ξέρετε ότι το σκάφος που είναι το πιο γνωστό στο στόλο μας αυτή τη στιγμή είναι αυτό που πηγαίνει να κάνει εξορίξεις ε, στη θάλασσα ε, για πετρέλαιο σε μεγάλα βάθη. Δεν νομίζω ότι με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να λύσουμε το πρόβλημα και εδώ υπάρχουν πολύ καλοί λόγοι για να να φαίνεται τόσο ελκυστική η γαλάζια οικονομία. Καλή και κάποιοι λιγότερο καλή. Έχουμε ένα πληθυσμό που αυξάνεται. Έχουμε έλλειψη φυσικών πόρων στη γη, στην ξηρά. Έχουμε οικονομική παγκοσμιοποίηση που εντείνεται και θα συνεχίσει να εντείνεται. Έχουμε μεταφορές εμπορευμάτων και όπως είπα έχουμε και τεχνολογικά μέσα που επιτρέπουν φοβερά κατορθώματα σε σχέση με κάποια χρόνια. Αυτά είναι τα θετικά. Όμω, κατά τη δική μου αντίληψη, εδώ προκύπτουν κάποιε υποχρεώσει, κάποιε επιτακτικέ ανάγκε. Πρώτα απ' όλα, να μην ξανακάνουμε στη θάλασσα αυτό που κάναμε στην ξηρά στη γη. Επίση, για αυτό το λόγο, να αλλάξουμε ε, μοντέλο εκμετάλλευση. Θα έπρεπε να ξεχάσουμε τελείω τον όρο μοντέλο εκμετάλλευση. Πρέπει να βρούμε ένα καινούριο όρο. Και γιατί. Γιατί στην γη, στην ξηρά, τι κάναμε. Κατασπαταλήσαμε διαπράξαμε σφάλματα που δεν ε, διορθώνονται, οικοκτονίες θα τις έλεγα, οικολογικές οικοκτονίες, εγκλήματα κατά του περιβάλλοντος, κατασπατάληση, κατασπατάληση φυσικών πόρων που δεν μπορούν να ανανεωθούν. Πρέπει να αλλάξουμε εντελώ λοιπόν μοντέλο, πρότυπο. Και εδώ θα συμφωνήσω με αυτό που προηγουμένω η Κλαρά Αγγιλέρα. Στην Ένωση θα πρέπει να προσπαθήσουμε να κάνουμε αυτό που ξεκινήσαμε στην Αλία και την μέγιστη απόδοση, ακόμη και αν δεν είναι η καλύτερη, ακόμη και αν βελτιώνεται. Ε, πρέπει να το πιστέψουμε παρόλα αυτά, ε, γιατί θα πρέπει από του φυσικού πόρου να παίρνουμε αυτό που μπορεί να, να παραχθεί. Δεν μπορούμε να επιτιθέμεθα στο κεφάλαιο των φυσικών πόρων και να παίρνουμε ό,τι μα ενδιαφέρει ε, και να μην ε, τραβάμε για να, όπως από ένα λογαριασμό για να χρησιμοποιήσω μια έκφραση των ε, καπιταλιστών. Θα πρέπει λοιπόν να αποφύγουμε τις βλαπερές συνέπειες για τα αποθέματα και τους φυσικούς πόρους εν γέννη. Χρειάζονται πολλά εδώ, αλλά δεν θέλω να μακρηγορήσω. Είναι δύο οι βασικές απαιτήσει. Πρώτα απ' όλα, να κοιτάξουμε την καλή διαχείριση των πόρων και των οικοσυστημάτων. Διότι δεν είναι δεδομένα αυτά, και εδώ θα συμφωνήσω με του πρόγραμμου ομιλητέ, και ναι, το θέμα των ελέγχων, το θέμα τη αστυνόμευση. Πρέπει να κοιτάμε ποιο κάνει τι. Συχνά δεν αρκεί η εμπιστοσύνη, δεν γεννάει έλεγχο. Ω προς την παραγωγή και την παραγωγή πλούτου, καθώς και την εκμετάλλευση των φυσικών πόρων, ο έλεγχο είναι ε, κέρια σημασία. Για να ολοκληρώσω, να πω, <clears throat> για να είμαστε αποτελεσματικοί και σοβαροί και να φτάσουμε στο τέρμα ε, των όσων λέμε, των υποχρεώσεων του δρόμου μας, θα πρέπει να βγούμε από τις αποκλειστικές οικονομικές ζώνες και την λογική των, οικονομικ... εθνικών εγωισμών. Θα πρέπει να αφήσουμε τα 10 και τα 12 μίλια και θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση επιτέλους να συνειδητοποιήσει ότι υπήρξε χερσόνησος, κατακαιρματισμένο ήπειρος και μια από τις πιο θαλάσσιες, τις ναυτικές ήπειρους. Μας περιβάλλει νερό, δεν είναι και λίγο αυτό για τα θεσμικά μας όργανα, κύριε Επίτροπε. Έχουμε μια γενική διεύθυνση που ασχολείται υποτίθεται μόνο με την Αλία, τη Μάρε. Εδώ στο Ευρωκοινοβούλιο έχουμε μια επιτροπή, την Επιτροπή Αλία, που υποτίθεται ότι ασχολείται με την Αλία. Αλλά έχουμε και τι θαλάσσιε μεταφορέ την Επιτροπή Μεταφορών, τέσπα, μην πολύ λόγο. Δεν θα σας τα πω όσα υπάρχουν, αλλά ακόμα δεν έχουμε συνέστηση, δεν έχουμε συνειδητοποιήσει πλήρω ότι η Ευρώπη είναι θαλάσσια και ναυτική. Τι θα γίνει λοιπόν με τη θαλάσσια κυβέρνηση, το είπα, και για να ολοκληρώσω, Πρόεδρε, δυο λόγια για την ανθρωπότητα. Να μην ξεχνάμε την ανθρωπότητα στους ωκεανούς και να μην ξεχνάμε κατά κύριο λόγο το δικαίωμα, μάλλον την υποχρέωση, το καθήκον της διάσωσης στη θάλασσα. Η διάσωση των, της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα είναι αρχή, αξία που ισχύει από αιώνες απαράβατη και τώρα την εγκαταλείπει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Thank you. And now uh, we have a couple of speakers. Uh, each one uh, I would like to ask to really stick to the... Θα ήθελα να σας παρακαλέσω να τηρείτε το πεντάλεπτό σας. Ο κύριος Βίτο Βερτέλιο από την Ένωση για τη Βιομάζα στην Ευρώπη. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ και ε, τους διοργανωτές για την πρόσκληση. Εγώ θα ήθελα να σας μιλήσω για τρία θέματα. Πρώτον, να σας εξηγήσω ε, τι είναι τα φύκια. Ποιο είναι το πρόβλημα ε, στην υγεία των ωκεανών και τι ρόλο μπορούν να παίξουν τα φύκια για να προσπαθήσουμε να λύσουμε το πρόβλημα. Τι είναι η βιομάζα από τα φύκη. Είναι μικροφύκη, πολύ μικροσκοπικά, που καλύπτουν ε, όλους τους ωκεανούς ε, και ε, με τη φωτοσύνθεσή τους ε, παράγουν οξυγόνο, όπως ακούσαμε. Αυτή τη μορφή έχουν. Είναι το ένα χιλιοστό του ενός χιλιοστού. Υπάρχουν πάρα πολλές ποικιλίε και είδη με διάφορα ονόματα. Αυτά είναι από τα πιο διεδομένα μικροφύκη στον πλανήτη. Ε, καλύπτει το 5% της φωτοσύνθεσης των ωκεανών. Και ποια είναι τα πολύ μικροσκοπικά φύκη. Είναι αυτά τα φύκη που βλέπετε εδώ, στις ακτές επίσης. Ε, ε, σας δείχνω μερικές φωτογραφίες. Αυθονούν στην Ευρώπη στην Ασία ε, καλλιεργούν αυτά τα φύκια. Στην Ευρώπη τα συλλέγουν από τους ωκεανούς, τις ε, Έχουν διαφορετικές δραστηριότητες ε, και ιδιότητες τα διάφορα φύκια. Μπορούν να παράγουν πολλοί σακχαρίτες, μπορούν να επεξεργάζονται σε βιολογικό καθαρισμό τα α, Αυτό το φύγι που σας δείχνω τώρα, το κόκκινο, αυθονούσε στην Πορτογαλία, στη χώρα μου, αλλά ε, υπερεκμεταλλεύτηκαν ε, αυτό το είδος ε, οι άνθρωποι και τώρα σχεδόν έχει εξαφανιστεί. Να σας πω δύο λόγια και για το πρόβλημα ποιο είναι. Της υγείας των ωκεανών ουσιαστικά από την μη βιώσιμη εκμετάλλευση των ωκεανών. Εδώ βλέπουμε σε αυτή τη διαφάνεια ότι δύο είναι τα βασικά προβλήματα. Το ένα είναι η ρήπανση και το δεύτερο είναι η υπεραλίευση. Η ρήπανση έχει πολλές εκφάνσεις και πτυχές. Ε, έχει υπερβολική η έκκληση διοξιδίου του άνθρακα ε, στην ατμόσφαιρα αλλάζει το κλίμα και αυτό προκαλεί πολλά προβλήματα στους ωκεανούς. Άλλο πρόβλημα είναι τα πλαστικά που αναφέρθηκαν για τη ρήπανση και η υπεραλίευση έχει σχέση με αυτά. Το θέμα των πλαστικών κατά την προσωπική μου άποψη είναι από τα βασικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε τώρα. Όχι τα μεγάλα πλαστικά αλλά τα πολύ μικροσκοπικά πλαστικά γιατί αυτά τα πλαστικά δεν προέρχονται μόνο από την αποσύνθεση των ίδιων των πλαστικών από τη διάσπαση, αλλά ε, και από ε, την πλήση όλων των ρούχων που χρησιμοποιούμε και εγώ τα χρησιμοποιώ που δεν είναι όλα βαμβακερά αλλά είναι συνθετικά. Κάθε φορά που πλένουμε ένα ρούχο συνθετικό, δηλαδή πλαστικό, απελευθερώνονται σωματίδια μικροσκοπικά πλαστικών και καταλήγουν στον ωκεανό. 6 με 9 εκατομμύρια τόνοι το χρόνο. Εκατομμύρια τόνοι. Αυτό είναι τεράστιο ε, ποσό. Και αυτά τα μικροπλαστικά για να διασπαστούν χρειάζονται χίλια χρόνια και δεν μπορούν να απομακρυνθούν με κανένα τρόπο από τους ωκεανούς. Είναι τόσο μικροσκοπικά, ε, ε, αυθονούν, είναι ε, παντού και τα τρώνε τα αμαλάκια, οι πολύ μικρές γαρίδες, τα ψάρια και περνάνε στην τροφική αλυσίδα και τελικά καταλήγουν και στον άνθρωπο. Αλλά ας είμαστε λίγο πιο θετικοί και αισιόδοξοι. Πώς μπορούν να συνεισφέρουν τα φύκη λοιπόν. Δύο είναι τα βασικά προβλήματα στον ωκεανό. Το ένα είναι τι βάζουμε, τι ρίχνουμε δηλαδή, τι πετάμε στους ωκεανούς και το άλλο είναι τι βγάζουμε από τους ωκεανούς. Τι ρίχνουμε εκεί. Ένα σωρό ε, χημικούς ε, και τι βγάζουμε με την υπεραλίευση ψάρια αλλά και, και θηλαστικά, δελφίνια, ε, ε και ε, μα, μαλάκια και οστρακοειδή, ε, πολύ μικρές γαρίδες, ακόμα και στην Αρκτική. Σε τρία επίπεδα είναι η δράση μας. Το πρώτο είναι η πρόληψη. Το σημαντικότερο είναι να τα σταματήσουμε όλα αυτά. Όχι απλώς να καθαρίσουμε τους ωκεανούς, με την πρόληψη να τα σταματήσουμε όλα αυτά και να έχουμε μια οικονομία πιο κυκλική, χωρίς πλαστικά, χωρίς διοξίδιο του άνθρακα και ε, μια δεσμευτική βιωσιμότητα και ε, πολύ δρακόντια φορολογία για οτιδήποτε ρηπαίνει τους ωκεανούς. Μετά, ενημέρωση. Κατά την άποψή μου είναι το σημαντικότερο. Οι πολίτες, αν δεν γνωρίζουν τι συμβαίνει, δεν πρόκειται να πιέσουν τους πολιτικούς και οι πολιτικοί θα δρανήσουν. Και τέλος, χρειάζεται να έχουμε ισόρροπη εκμετάλλευση των θαλασσών και των ωκεανών. Ε, με την υπερεκμετάλλευση δεν προστατεύεται ο ωκεανός. Τι μπορούν λοιπόν τα φύκη να κάνουν για όλα αυτά τα πράγματα. Τέσσερα κυρίως. Τα δύο πρώτα είναι ότι μπορούν να αντικαταστήσουν τις ε, ηχθειοτροφές, στις ηχθειοκαλλιέργειες. Στην ιδιατοκαλλιέργεια χρησιμοποιούμε 7 εκατομμύρια τόνους το χρόνο ηχθιέλαια και ηχθιάλευρα και 200 εκατομμύρια τόνους ε, ε, αλεύρια από σόγια και σογέλαιο. Μπορούν τα φύκια αυτό να το αντικαταστήσουν όταν παραγόνται σε πολύ μεγάλη κλίμακα. Και έτσι ε, θα αλλιεύουμε λιγότερα ψαράκια για να τα κάνουμε ηχθιάλευρα. Και έτσι θα σωθούν και δάση στη ξηρά. Ε, μπορώ να σας δείξω πολλές εφαρμογές στην επόμενη διαφάνεια. Να σας πω ότι τα φύκη μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν ε, για ε, επιλεκτική αποκατάσταση βιολογική. Δηλαδή, τα φύκια μπορεί να είναι φορείς βακτηρίων που διασπούν τα πλαστικά. Επίσης, άλλη ιδιότητα να είναι η λίπανση των ωκεανών, όπου έχουμε νεκρές ζώνες χωρίς οξυγόνο, μπορούν τα φύκη να δημιουργήσουν ζώνες που να παράγεται οξυγόνο και αυτό να αλλάξει ριζικά το θέμα της κλιματικής αλλαγής. Και τέλος είναι οκτώ οι βασικές εφαρμογές των φυκών και των πολύ μικροσκοπικών και των κανονικών φυκιών που φυτρώνουν στη θάλασσα. Ε, τροφές, ζωοτροφές, ε, λιπάσματα, χημικά, καλλιντικά κλπ. Και η Ευρώπη είναι ηγέτης εκεί. Υπάρχουν πολλά ερευνητικά προγράμματα στην Ευρώπη σε όλους αυτούς τους τομείς. Αυτά και τελείωσα και σας ευχαριστώ. Thank you. And now, uh, σας ευχαριστώ και τώρα η κυρία Ασίνα, διευθύντρια του Policy Office του WWF για πέντε λεπτά παρακαλώ. Θα προσπαθήσω να τα καταφέρω και ευχαριστώ και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την οργάνωση της διάσκεψης αυτής. Χαίρομαι Εκπροσωπώ εδώ την οργανώσή μου που έχει συνεισφέρει στην ανάπτυξη της αρχής, των αρχών μάλλον, της βιώσιμης γαλάζιας οικονομίας. Κάποιοι είπαν ε, ότι ο ωκεανός μοιάζει σαν το και εκτιμήσαμε ότι υπάρχει πολύ μεγάλη αξία στην ωκεανή οικονομία, περίπου 24 τρισεκατομμύρια δολάρια, τα οποία μπορεί να, μεταφραστούν σε κέρδη περίπου σε 2,5 τρισεκατομμύρια δολάρια χωρίς να μιλήσουμε για όλα τα άλλη ωφέλη, το οξυγόνο, τα τρόφιμα, αλλά αποτελεί και ε, αναχέτηση, παράγοντα αναχέτησης κλιματικής απειλής. Επίσης, ε, η οικονομία του ανακαινού αναμένεται να διπλασιαστεί μέχρι το 2030 κατά μέγεθος και ε, δημιουργεί ένα προηγούμενο για τις μεταφορές, τη βιοτεχνολογία, την ενέργεια. Ε, πέρα από ότι εμείς μα οργανώσει ενδιαφερόμαστε για τη βιοπικιλότητα, όταν βλέπουμε τους δείκτες της υγείας των ωκεανών, δεν οδεύουν προς τη σωστή κατεύθυνση, αντιθέτως ε, κινούνται προς τη λανθασμένη κατεύθυνση. Περίπου το ένα τμήμα, το ένα τρίτο συγγνώμη, των ελευτικών επελευμάτων ε, ε, οι, λιμόνες, ε, συγγνώμη, η μαγκρόβια βλάστηση ε, αποψηλώνονται δύο-τρεις φορές ε, ταχύτερα από τα τροπικά δάση. Μιλάμε για τα τοξικά, τα πλαστικά και την κλιματική αλλαγή. Όλα αυτά έχουν πολύ σοβαρό αντίκτυπο στις παράκτιες περιοχές, αλλά και για την οξύνηση των πιο κρυών υδάτων έχουν αντίκτυπα, αντίκτυπο στην τροφική αλυσίδα. Και κάτι ακόμη που αφορά τον την οργάνωσή μου αφορά την ελεύκανση των κοραλιών γιατί είδαμε πριν ε, δύο χρόνια το πιο σοβαρό περιστατικό λεύκαρση των κορελιών. Χάσαμε σχεδόν το ίμιση των κοραλιογενών υφάλων και αν συνεχίσουμε με την ε, σημερινή τάση θα τους χάσουμε όλους τους υφάλους μέχρι το 2050 και όχι απλώς ε, χάνουμε ένα πολύ όμορφο είδος αλλά έχει αντίκτυπο αυτό σε εκατομμύρια ανθρώπους από το οποίο εξαρτώνται για το εισόδημά τους και για την προστασία των παράκτων περιοχών τους. Αν έχουμε καλή διαχείριση των ωκεανών, τότε θα συνεισφέρει στο να πετύχουμε όλου του 17 στόχου τη βιώσιμη ανάπτυξη και αυτά είναι καλά νέα. Αλλά για να επανέλθω σε ό,τι είπε προηγούμενο ομιλητή, οι φιλοδοξίε μα για την οικονομική ανάπτυξη εξαρτώνται από υγιή οικοσυστήματα και τι υπηρεσίε που προσφέρουν. Για να τα πούμε πολύ απλά λοιπόν δεν θα έπρεπε να μιλάμε για τη φιλοδοξία μα για την ε, γαλάζια ανάπτυξη, αλλά θα πρέπει να μιλάμε για την ανάγκη ελαχιστοποίηση του κινδύνου και να δημιουργήσουμε ανθεκτικότητα στου ωκεανού ε, εν ώψη της κλιματική απειλή. Αυτό απαιτεί να προστατεύσουμε πολλά από αυτά τα οικοσυστήματα πρέπει από το να σκεφτούμε πώς θα τα εκμεταλλευτούμε και να λάβουμε υπόψη τα όρια του πλανήτη γιατί ξέρουμε ότι έχουμε μόνο ένα πλανήτη και αυτό θα απαιτήσει σημαντικές επενδύσεις προκειμένου να αποκαταστήσουμε αυτό το φυσικό κεφάλαιο που είναι υποπηλή σήμερα. Θα πρέπει να θεωρηθεί αυτό Μέρο όλη ε, τη επιχειρηματική πρόταση. Είμαστε λοιπόν σε σημαντικό σταυροδρόμι και αναφέρθηκε αυτό και από νεότερου συναδέλφους. Ε, από την ε, μία πλευρά έχουμε πολιτέ που ζητάνε όλο και περισσότερο δράση και από την άλλη έχουμε τι δημόσιε πολιτικέ και είναι ένα βήμα μπροστά η Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί έχει ήδη τα νομοθετικά εργαλεία για τη βιώσιμη γαλάζια οικονομία αλλά τώρα πρέπει να εφαρμόσουμε αυτά τα εργαλεία και θέλω να αναφέρω τρία. Το πρώτο αφορά τη στόχους της κοινή ελευθερικής πολιτικής για την επίτευξη βιώσιμης αλίας μέχρι το 2020, αλλά και την οδηγία πλαίσιο για ε, την θαλάσσια στρατηγική 2020 και αυτό πολύ σύντομα. Και μια άλλη πολιτική σημαντική είναι η σύμβαση για την βιοπικιλότητα, ο στόχος 11 που καλεί για την προστασία τουλάχιστον 10% ε, των ε, παράκτιων και θαλάσσιων περιοχών. Λεχθέντων ε, αυτών, νομίζω ότι πρέπει να ξαναπούμε, τώρα καλούμε για δράση. Το 2020 θα κάνουμε μία αποτίμηση πολλών διεθνών συμφωνιών, της Συμφωνίας των Παρισίων, των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης και τη Σύμβαση για την Βιοτοπική Βιοπικιλότητα, τη CBD. Και γι' αυτό καλούμε για μια νέα όθηση για τη φύση, μια νέα συμφωνία, ένα νέο deal για τη φύση και για τους ωκεανούς και τη βιοπικιλότητα. Πρέπει να ενταχθούν πολύ περισσότερο στο επίκεντρο του πολιτικού θεματολογίου. Και θα κλείσω με τα τρία μήνυματά μου και θα στήσω από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Καταρχήν, να απαντήσει την παγκοσμία κλίση για βιώσιμε επενδύσει και ανάπτυξη στην ε, παγκοσμία γαλάζια οικονομία. Δεύτερον, και παγκοσμίω και εσωτερικά να προωθήσει τη βιώσιμη ελεία και την κυκλική οικονομία και να προστατεύσει τρίτον την αρθεκτικότητα των ωκεανών εγκαίρως για την προθεσμία του 2020. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ και για την τήρηση του χρόνου. Ο κύριος Ζανεμιγκρούτσε, πάλι για πέντε λεπτά. Από το Energy Europe. Ευχαριστώ πολύ κύριε Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα σε όλους, Επίτροπε, κύριοι βουλευτές, συνάδελφοι. Η δική μας οργάνωση εκπροσωπεί την ενέργεια στους ωκεανούς. Θα ήθελα αυτή τη στιγμή να επικεντρωθώ στην Παλήρια και στα παλιριακά κύματα. Εδώ λοιπόν στις εικόνες βλέπετε τι συμβαίνει Πατήστε το ένα παρακαλώ. Μπορεί να ρωτηθείτε. Τι τους χρειαζόμαστε, τους, τι, τι χρειαζόμαστε την ενέργεια από τους ωκεανούς. Έχω μια διπλή απάντηση. Η πρώτη είναι το κλίμα και η άλλη η μηχανική ανάπτυξη. Το κλίμα προφανώς, διότι ξέρουμε ότι ως το 2050 δεν μπορούμε να ε, έχουμε την παραμικρή εκπομπή άνθρακα πλέον για την παραγωγή ηλεκτρικού. Πρέπει να υπάρχει ανανεώσιμη παραγωγή. Εάν δείτε την έκθεση του IPPC, τα σενάρια τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. τα περισσότερα πιστεύουν ότι πρέπει να φτάσουμε το στόχο της ανανεώσιμης ε, ενέργειας μέχρι το 2050 κατά 100%. Για να γίνει αυτό θα πρέπει να είναι βιώσιμη και η ζήτηση και η προσφορά. Για να εξορροπήσουμε τις δύο αυτές ε, διαστάσεις χρειάζεται η κατάλληλη παραγωγή ενέργειας και αποτελεσματικότητα στην ενέργεια, απόδοση στην ενέργεια μάλλον και η σωστή αποθήκευση και γι' αυτό χρειαζόμαστε καταπληρωτικά κύματα. Γιατί διότι παράγουμε πολύ διαφορετικό ρυθμό από τη ολική και η ηλιακή ηλεκτρική ενέργεια. Θα μπορούσαμε να ελαφρύνουμε τα σχετικά συστήματα. Μέχρι το 2050 μπορούμε να φτάσουμε 10% της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας από τα παλιωτικά κύματα των ωκεανών. Το δεύτερο έχει να κάνει με τη βιομηχανική ανάπτυξη. Η ενέργεια των ωκεανών. Α, να το λέει. Η ενέργεια των ωκεανών σημαίνει και επενδύσει. Και κέρδο. Η Δανία, η Γερμανία έχουν ήδη ωφεληθεί στην διεθνή αγορά, αξιοποιώντα του ωκεανού. Αυτό μπορεί να γίνει και σε άλλε περιοχέ, σε άλλε χώρε τη Ευρώπη που είναι παραθαλάσσιες μπορούμε να δημιουργήσουμε 400.000 θέσει εργασία στην Ευρώπη και αρκετέ και εκτό. Έχουμε πετύχει αρκετά στι διάφορε ακτέ. Αυτά που δείχνουμε προ τη είναι ακριβά ίσω, Αλλά έχουμε κατεβάσει το κόστο για την νεολική και την ηλιακή ούτω ή άλλω και ανάλογο μπορούμε να κάνουμε, κάτι ανάλογο μπορούμε να κάνουμε για, τη, για τους ωκεανούς. Λίγο τσιμέντο, λίγο μπετόν, ε, κάποια καλώδια και κάτι άλλα εξαρτήματα χρειαζόμαστε και μετά μπορούμε με απλά μηχανήματα να αρχίσουμε να παράγουμε. Η πράσινη ανάπτυξη χρησιμοποιείται ήδη στην ε, ηλιακή και την αιωλική. Θέλουμε το ίδιο να γίνει και στους ωκεανούς λοιπόν. Ε, το γαλάζιο κατά κάποιο τρόπο είναι το νέο πράσινο που θα έλεγε κάποιος ε, όπως και το όνομα της σειράς εδώ λοιπόν θα πρέπει να κάνουμε κάτι και γι' αυτό, για τον περιορισμένο αντίκτυπο ανάλογα με το ποια σκοπιά υιοθετήσει κανείς και το τι αντικτύπους βλέπει στο τοπικό περιβάλλον. Έχουμε τη δυνατότητα να ε, ε, ενεργοποιηθούμε σε περιοχές όπου υπάρχουν ισχυρά ρεύματα. Εκεί όπου υπάρχει λιγότερη βιοπικιλότητα, γιατί ο πυθμένης της θάλασσας είναι βράχια, σκληρά βράχια. Ε, συμπαγή. Αυτό που χρειαζόμαστε λοιπόν είναι περισσότεροι δακτύλοι, περισσότεροι περισσότερες άγκυρες που να μην καταστρέφουν το θαλάσσιο πυθμένα. Εδώ λοιπόν πρέπει να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε καλύτερα για την παραγωγή ενέργειας. Ε, για τα θηλαστικά, ε, για μια σειρά από ενέργειες στη θάλασσα, ειδικά για τις φώκες ας πούμε, και γιατί για την ώρα δεν έχουμε παρατηρήσει να υπάρχουν ε, άλλου είδους προβλήματα μεταξύ τη προστασία των ειδών. Εδώ λοιπόν το νέο πράσινο είναι το γαλάζιο. Θέλουμε να δούμε πώς μπορούμε να πάμε ως εκεί με τρόπο βιώσιμο και για την αίμα που ζητά να έρθει ο ιδιωτικό τομέα και να αναλάβει πρωτοβουλίες και να επενδύσει, τα ξέρει καλά, φαντάζομαι, αλλά οι επενδυτέ χρειάζονται δύο πράγματα για να επενδύσουν σε νέε τεχνολογίε. Χρειάζονται προβλεψιμότητα και χρειάζονται και κίνητρα. Σας ευχαριστώ λοιπόν εδώ για την πρόσκληση. Σας ευχαριστώ κύριε Βέλα, κύριε Μοέδα, για τα πέντε χρόνια σκληρής δουλειά πολιτικού και οικονομική ενίσχυση. Χωρί εσά κάποιε από αυτέ τι διαφάνειε, κάποιε από αυτέ τι τεχνολογικέ λύσει, δεν θα έπλεαν σήμερα στους ωκεανούς όπως σήμερα. Έχουμε πάρει λίγη χρηματοδότηση από τον ορίζοντα 2020. Κάποιες από τις συσκευέ αυτές δεν θα υπήρχαν στη θάλασσα, δεν θα τις είχαμε τρέξει εάν δεν είχατε βοηθήσει κι εσείς. Έκλεισε ε, για δράση, προ ε, για δράση προς τα κράτη-μέλη λοιπόν εδώ, ιδίω στη χώρα των Βάσκων ας πούμε, που έχει πετύχει ιστορικά βήματα πρώτα. Ε, σε εθνικό επίπεδο χρειαζόμαστε προβλεψιμότητα στην αγορά ε, και προβολή και κάτι που να προσελκύσει του επενδυτέ. Δεν θα επενδύσουν αλλιώ οι επενδυτέ σε ένα καπιταλιστικό κόσμο χωρί αυτά τα δύο στοιχεία. Εάν είναι κανεί λοιπόν εκπρόσωπο κάτω μέλου, βουλευτή από κάτω μέλου, παρατηρούμε, δείτε τι γίνεται με την ενέργεια ε, και τι γίνεται με την τεχνολογία που χρησιμοποιείτε. Αν δεν το κάνετε για τις βιομηχανίες, κάντε το για τις κοινότητες που ζουν σε παράκτητες περιοχές. Έχουν υποφεληθεί ε, πάρα πολύ από αυτό το είδος την επιχειρηματική δράση, το ίδιο και θα υποφεληθούν από την παραγωγή ενέργειας. Ευχαριστούμε λοιπόν πολύ. Εάν σας ενδιαφέρουν όσα κάνουμε, κοιτά, ψάξτε μας στο Google. Θα είναι χαρά μας να συνεργαστούμε τις επόμενες δεκαετίες για τα θέματα αυτά και την παραγωγή καθαρής ενέργειας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Τρουέ. Και τώρα θα παρακαλούσα τον τελευταίο ομιλητή να πάρει το λόγο, Κρίστοφ Τούτκατ, Γενικός Γραμματέας της c Europe. Thank you, Chairman. Um, dear Commissioner. Ευχαριστώ. Κύριε Πίτροπε, κύριε Μάισνερ, Κυρίε και κύριοι, καλησπέρα. Καταρχήν, ε, θα ήθελα να ευχαριστήσω του διοργανωτέ τη σημερινή συνεδρίαση που κάλεσαν ε, το ΣΥΓΙΟΡΟΠΑ. Για όσου δεν μα ξέρετε, είναι οργάνωση που εκπροσωπεί τα συμφέροντα των ναυπηγείων και όσους ε, κατασκευάζουν εξοπλισμό συλλογικά. Είμαστε πάνω από 8.000 εταιρείε σε ευρωπαϊκό πλαίσιο και εκπροσωπούμε τον ευρωπαϊκό τομέα τεχνολογία. Τώρα, τι κάνει ε, μια τέτοια οργάνωση σε μια σύνοδο για τους ωκεανούς. Θα προσπαθήσω να σας εξηγήσω ότι είναι καταρχήν η συντήρηση, η μετατροπή ε, και η επισκευή του εξοπλισμού πολύπλοκων ε, πλατφόρμων offshore και πλέον και εξακολουθούμε να έχουμε στην Ευρώπη μια παγκόσμια ηγετική θέση και είμαστε περήφανοι, αλλά πάμε και λίγο παραπέρα. Εξετάζουμε περισσότερο την τεχνολογία και τις υποδομές που είναι κατάλληλες για τις ε, ε, δραστηριότητες της γαλλικής οικονομίας. Αν δείτε τα κρουαζερόπλια, πιστεύουμε ότι είναι ένα αυτό πολύ σημαντικό ε, τμήμα των δραστηριοτήτων ε, και κατασκευάζονται σε ευρωπαϊκό πλαίσιο. Έτσι λοιπόν, ο τομέα μα ε, έχει στην καρδιά του του ωκεανού και τι θάλασσε και θέλει να συνεισφέρει σε βιώσιμη γαλάζια οικονομία και να μειώσει την πίεση που υπάρχει στους ωκεανούς. Και αυτό δεν το κάνουμε μόνο μας, το κάνουμε με τους συναδέλφους, με την Waterboard Technology Platform. Αυτή η πλατφόρμα είναι ε, μια νέα στρατηγική ε, ερευνητική ατζέντα και ε, εκεί καλύπτει όχι μόνο τις κλασικές μεταφορές θα αναφέρω πιο συγκεκριμένα. Καταρχήν, τις θαλάσσιες μεταφορές. Αυτό σημαίνει τα παντοπόρα πλοία, αλλά και την εσωτερική ναυσιπλοεία. Εδώ θέλουμε ένα καθαρό ε, τρόπο μεταφορών. Θέλουμε μέχρι το 2030 να φτιάξουμε νέα ποντοπόρα πλοία αλλά και εσωτερική ναυσιπλοεία ε, με μηδενικέ εκπομπέ. Ενώ για τα άλλα σκάφη θέλουμε μείωση 50% των εκπομπών ενώ θα πλέον στη θάλασσα. Και μέχρι το 2050 πιστεύουμε ότι μπορούμε για κάθε πλοίο να έχουμε μηδενικέ εκπομπέ. Και όταν μιλάμε για μηδενικέ εκπομπέ, δεν μιλάμε μόνο για τη μείωση των εκπομπών στην ατμόσφαιρα και των αερίων του θερμοκηπίου, αλλά μιλάμε και για τη μείωση τη ρήπανση θάλασσα και τη συγχωρήπανση. Και με αυτή την ε, φιλοδοξία ε, θέλουμε να πάμε πέρα από αυτά που συζητάτε, συζητώνται σήμερα στο πλαίσιο ε, του Διεθνούς Οργανισμού Ναυσιπλοείας ε, στο Λονδίνο, αλλά πέρα από το να έχουμε πλωτές μεταφορές, ε, καθαρές και πράσινες, θέλουμε να δούμε και τις γαλάζιες δραστηριότητες, τις δραστηριότητες γαλάζιας οικονομίας. Προηγούμενη ομιλήτρια αναφέρεται, προηγούμενος ομιλητής, συγγνώμη, αναφέρθηκε σε αυτό, οπότε δεν θα αναφερθώ και εγώ αλλά θα επικεντρωθώ σε άλλα πράγματα. Καταρχήν, θέλουμε να προωθήσουμε την προστασία των ωκεανών και των εσωτερικών πλωτών οδών. Πιστεύουμε ότι μέχρι το 2030 θα πρέπει η Ευρώπη να έχει πλήρη ε, ολοκληρωμένη ένα πλήρως ολοκληρωμένο σύστημα ε, παρακολούθησης ε, των ωκεανών και των θαλασσών και να έχουμε μία ολιστική εικόνα όλων των πλωτών επιχειρήσεων και έτσι θα μπορούμε να έχουμε επιχειρήσεις για απορρίμμαση από τα πλαστικά. Επίσης θέλουμε να διευκολύνουμε ε, στις offshore ε, πλατφόρμες ε, να αναπτύξουμε πολλαπλά συστήματα για να προστατεύσουμε τους εργαζομένους στις, παράκτης, στις πλατφόρμες να έχουμε καλές συνθήκες διαβίωσης στη θάλασσα. Ε, και με τέτοιους συνδυασμούς με υπεράκτιες πλατφόρμες ε, θέλουμε να παράγουμε στην Ευρώπη τα πρώτα πλωτά νησιά ε, για Κάποιε ε, βιομηχανικές δραστηριότητες ή ψυχακικές δραστηριότητες και κατοικία μέχρι το 2050. Ε, βέβαια πρέπει να πληρούνται πολλές προποθέσει. και καταρχήν και το έφεραν και κάποιοι προηγούμενοι ομιλητέ, η ανάγκη για σημαντικέ επενδύσεις ε, στην έρευνα, στην ανάπτυξη και στην κοινοτομία και στο πλαίσιο του ορίζων Ευρώπη αλλά και εκτό του πλαισίου Horizon Ευρώπη. Σήμερα ο τομέα τη θαλάσσια τεχνολογία επενδύει το 10% σε δραστηριότητε έρευνα και ανάπτυξη ε, και είναι ένα από του πρωτοπόρου σε βιομηχανική έρευνα και ανάπτυξη. Αλλά αν θέλουμε να αναπτύξουμε το δυναμικό τη γαλάζια ε, ανάπτυξη ε, πλήρω και θέλουμε καθαρέ θαλάσσιε μεταφορέ, σίγουρα χρειάζονται περισσότερε επενδύσει σε έρευνα και ανάπτυξη. Δεύτερον, η εισαγωγή νέων τεχνολογιών και νέων ενιών θα πρέπει να υποστηρίζονται πλήρω με κατάλληλε πολιτικέ και κανονισμού. Αυτά είναι σημαντικά σε ευρωπαϊκό πλαίσιο συγκεκριμένα, γιατί πιστεύουμε ότι αυτό μπορεί να μας βοηθήσει για να είμαστε καινοτόμοι και το να, είμαι είμαστε καινοτόμοι σε ευρωπαϊκό πλαίσιο σημαίνει να είμαστε ανταγωνιστικοί σε παγκόσμιο κλίμακα. Τρίπον, λοιπόν, υπάρχει ανάγκη να υπάρχει ευκολότερη πρόσβαση στην ευρωπαϊκή χρηματοδότηση κυρίως ε, για ε, κεφαλικές επενδύσεις ε, και, και επενδύσεις με ένταση κινδύνου. Θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται καινοτόμα πλοία και πλατφόρμες και για δραστηριότητες γαλάζιας ανάπτυξης. Τέταρτον, ο κλάδος θα πρέπει να απασχολεί νέους με ενθουσιώδη κίνητρα και ε, με υψηλά προσόντα για να παράγουν καινοτόμες τεχνολογίες και να μπορούν να προσαρμοστούν σε έναν κόσμο τεχνολογικό που αλλάζει γρήγορα. Και τέλος, για τον ευρωπαϊκό ε, τομέα τεχνολογία στη θάλασσα, χρειαζόμαστε μια στρατηγική που την αποκαλούμε leadership strategy. Αυτό θα μας επιτρέψει να διατηρήσουμε την παγκόσμια ανταγωνιστικότητά μας ε, στον ε, παρασκευή, στην κατασκευή ε, του εξοπλισμού αλλά και την αφήγηση πλοίων και θα πρέπει να ωφεληθεί όχι μόνο ο τομέας αλλά και όλη η πλατική κοινότητα όπως και οι δραστηριότητες της γαλάζιας ανάπτυξης. Έτσι λοιπόν, ε, το μήνυμά μου με δύο λόγια είναι ότι θέλουμε γαλάζια ανάπτυξη και για τα ναυπηγεία. Είναι πολύ σημαντικό στοιχείο αυτό, είναι πολύ σημαντικό και για τις μελλοντικέ γενιές και για τον πλανήτη και θέλουμε να βάλουμε τα δυνατά μας να αναλάβουμε και τη δική μας ευθύνη προς αυτή την κατεύθυνση. Ευχαριστώ. Thank you, Mr. Ευχαριστώ πολύ. Εδώ ολοκληρώνεται το τελευταίο πάνελ υπαριθμών 3. Ξέρω ότι Ορισμένοι είναι έτοιμοι να κάνουν ερωτήσεις, αλλά με ενημέρωσαν ότι δεν μπορούμε να έχουμε ερωταπαντήσεις για τον απλούστατο λόγο ότι σε λίγο μας τελειώνει η διερμηνία. Και βεβαίως θέλετε να ακούσετε και το κλείσιμο και σας παρακαλώ να δείξετε κατανόηση. Σας ευχαριστώ γι' αυτό.